All Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα είναι αν έχουμε καμία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν νομίζω να έχουμε. Κρίνεται η ημερήσια διάταξη. Να περάσουμε λοιπόν σε μια σύντομη έκθεση τη συνεδρίαση των συντονιστών εχθέ το απόγευμα. Έληξα μια σειρά από αποφάσεις που επιβεβαιώνουν ε, την σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα πάει στην Ιταλία το Μάρτιο. Οι πράσινοι υποστηρίζουν ε, το αίτημα να χρησιμοποιήσει το Eurosember στο ημικύκλιο για την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Επιχειρήσεων κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2014 και θα γίνει μια αξιολόγηση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ε, μια προστιθέμενη αξία από τους Πρασίνους και καλούνται οι πολιτικές ομάδες ε, για ε, να προαρουσιάσουν ιδέες για εργαστήρια, μελέτες και το καθεξής. Ζητήθηκε από την Προεδρία να συντάξει μια επιστολή ε, μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας για να καθορίσουμε τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας για τον προϋπολογισμό του 2015. Επίσης, ε, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας ε, ζητήθηκε από την Προεδρία να συζητήσει το ζήτημα της συμφωνίας με το Μαρόκο και συμφωνήθηκε να αναβληθεί η απόφαση για την ανάθεση της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας ε, για την ε, σταθερότητα ε, των αγορών μετά του σύστημα εμπορίας εκπομπών, διότι εκκρεμεί η συνομιλία της Προέδρου με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνήθηκε να το ξανασυζητήσουν οι συντονιστές στην επόμενη του συνεδρίαση. Υπάρχει κάποια ερώτηση από αυτού? Η σιωπή σας εκλαμβάνετε ως συνένεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση για την κοινή επιχείρηση Shift to Rail, έκθεση της κυρίας ε, Αντρές Μπαρέα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή, όπως γνωρίζετε, είναι τμήμα ενός ε, πακέτου το οποίο ήρθε με κάποια καθυστέρηση και η επιχείρηση φαίνεται να έχει λίγο ε, μια κάποια στασιμότητα σε σχέση με το θέμα των σιδηροδρόμων. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες προσπάθειες και ήταν ικανοποιητικές, τώρα έγινε μια αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και έχουμε εντοπίσει και κάποια σημεία τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν λειτουργεί και τόσο αποτελεσματικά το σύστημα. Ε, λόγω έλλειψη συντονισμού, λόγω αλληλοεπικαλύψεων και δεν έχει υπάρξει και ιδιωτικό ε, κεφάλαιο ω επένδυση και δεν υπάρχει και συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη δέσμη λοιπόν αυτών μέτρων θα πρέπει να κάνουμε ε, κάποιες προσπάθειες, να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση, να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντο, να μειώσουμε λίγο το κόστος ε, ω προ τη συνολική ζωή των μεταφορών, της υποδομές, ε, για το τροχαίο υλικό, ε, αύξηση των δυνατοτήτων, ε, το τι χρησιμοποιείται και φυσικά να υπάρχει και μια κάποια αξιοπιστία και ασφάλεια για τους σιδηροδρόμους. Το Shift to Rail mm αναπτύσσει ένα master plus, plan ε, προτεραιότητας σε έρευνα και βασίζεται σε πέντε βασικά στοιχεία τα οποία είναι ουσιώδη η ποιότητα των υπηρεσιών, βελτίωση των υπηρεσιών, βελτίωση ε, της ασφάλειας, βελτίωση των εισιδημάτων, καλύτερη διαχείριση, έλεγχη της κίνησης, καλύτερες υποδομές, καλύτερη ασφάλεια και σαφήνεια, ε, αρνητικές συνέπειες, να αποφύγουμε τις παρενέργειες ε, ε, της εφιούς συντήρησης, να υπάρχει επικαιροποίηση του συστήματος των εισιτηρίων, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για το πώς ακριβώς μπορεί να γίνει ένα ταξίδι και να βελτιωθούν και τα θέματα της εφοδιαστικής. <clears throat> Διαπιστώσαμε διάφορες δυνατότητες Παρουσιάσαμε και τροπολογία για την συμμετοχή και τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις στο σχέδιο αυτό, αρκεί να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. 30 ε, εκατομμύρια ευρώ και 5 χρόνια δέσμευση για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επίσης για τους διαχειριστές των υποδομών. Ο προπολογισμό ο οποίος ε, υπάρχει είναι ε, της τάξης των 220 εκατομμυρίων, περιορισμένος προϋπολογισμός και η κατανομή κατά την άποψή μας δεν είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε ε, να είναι, γι' αυτό ακριβώς και υποβάλαμε σχετική τροπολογία. Ε, θα πρέπει η, το 40% να είναι από τις ιδρυτικές εταιρείες, το 30% από τους εταίρους και από εκεί και πέρα για τις συμπράξεις έχουμε ένα υπόλοιπο 30%. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και για τις ανοιχτές υποβολές προσφορών θα πρέπει να υπάρχει και πάλι μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Θα πρέπει όλα να τα βασίσουμε στη σωστή διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικό μεταξύ της ε, Επιτροπής ε, των ε, Συνεταίρων και των Ιδρυτικών Μελών. Επίσης, θα πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα βάση ανοιχτών μειοδοτικών διαγωνισμών και να τονίσουμε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των του Οργανισμού Σιδηροδρόμων ως δημόσια αρχή που ε, είναι αρμόδια για τα όσα συμβαίνουν. Ε, η συμμετοχή όλων μας φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της αγοράς. Υπάρχουν και παραδείγματα επιτυχίας στον τομέα αυτό, υπάρχουν κάποιες τεχνολογικές πρωτοβουλίες, κάποιες ε, κοινέ επιχειρήσεις και σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Shift to Rail διότι υπάρχει ένα άνοιγμα και προσφέρονται δυνατότητες για όλους όσους ε, πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και μεγαλύτερη εκπροσώπηση και να έχουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποβάλαμε μια σειρά από τροπολογίες οι οποίες ε, θα ε, μας φέρουν εκεί που επιθυμούμε, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή των κατάλληλων ευτεριών, αλλά κυρίως η ευελιξία και η δυνατότητα να γίνεται χρηστή διαχείριση μιας ε, κοινή επιχείρησης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές η έκθεση που παρουσιάσαμε. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαρέλη, ο Πρόεδρος. Και τώρα, οι σκιώδεις ιδέες έχουν το λόγο. Κυρία Καρβάλιο, νομίζω εσείς θα μιλήσετε εκ μέρους του κύριου Ντί. Έχετε το λόγο. Καλημέρα πρόεδρε και συνάδελφοι. Ο κύριος Ντί ζητεί συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί γιατί είχε κάποια υποχρέωση οικογενειακή. Οπότε μου ζήτησε να σας διαβιβάσω αυτά που έχει να πει πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο συζητούμε σε σχέση με το Horizon 2020, γιατί έτσι πρόκειται να τονωθεί η δυνατότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Έχουμε αυτές τις επιμέρους ε, πρωτοβουλίες, πρόκειται για συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, πρόκειται για ένα πρότυπο μοναδικό και επίσης πετυχημένο. Το Shift to Rail, το οποίο συζητούμε τώρα, είναι μια καινούργια υπόθεση και το ΕΛΚ την στηρίζει. Ο κύριο Οντή θέλει να συγχαρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους όσοι έχουν εμπλακεί στην προετοιμασία αυτής της πρότασης και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας της Γιούνης ε, όλοι όσοι συνεργάστηκαν. Η πρόταση κανονισμού είναι πραγματικά αξιόλογη και ο κύριος Σοντή θα ήθελα να σας τονίσει ότι είναι υπέρ των οριζοντίων τροπολογιών που αφορούν τις επιμέρους τροπολογίες την απαλλαγή σε σχέση με το Horizon 2020, την ενδιάμεση αξιολόγηση κλπ. Όμως, όσον αφορά αυτή την περικοπή του 5% εδώ ακόμα επιφυλάσσεται. Το shift to rail συζητήθηκε και προετοιμάστηκε με, αφού ψηφίστηκε το Horizon 2020 και αφού συζητήθηκε ο προπολογισμό. Ο προπολογισμό, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη ε, έχει υποστεί αυτή την ε, περικοπή των 70 δις. Το 5% που θέλουν να προκόψουν και άλλο θα θεωρηθεί ότι αποτελεί έλλειψη στήριξης από δική μας πλευρά από την βιομηχανία. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ιδιορυθμίες στο Shift Rail και η έρευνα και η καινοτομία της ε, βιομηχανίας μας οδηγεί σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η βιομηχανία δεν πρόκειται να ζητήσουν παραπάνω πόρους από το ορίζον 2020 για το ζήτημα αυτό που συζητούμε. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες του, ο κύριος Οντή προβληματίζεται όσον αφορά αυτά τα περί ιδρυτικών τελεχών και τα περί κατανομής. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην ταράξουμε την ισορροπία πρέπει να ε, τα λάβει αυτά υπόψη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι. Α προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε πριν τον ε, Απριλίο. Ίσως η συγκήτρια μπορεί να προχωρήσει επί τη βάση του δικού της ε, χρονοδιαγράμματος. Ο κύριος ότι θεωρεί ότι το ζήτημα των ε, ιδρυτικών μελών, των άλλων μελών, των εταίρων, θα πρέπει να, ε, θα πρέπει να ανακοινηθούν στο επίπεδο της βιομηχανίας και όχι σε επίπεδο πολιτικό, εδώ δηλαδή. Ελπίζουμε για τις τροπολογίες μας ότι θα στηρίξετε ό,τι έχουμε υποβάλει, κύριε Αντρές και οι άλλες και Έχουν δεσμευθεί 30 εκατομμύρια για όλη τη διάρκεια που θα τρέχει το Shift Rail και τα συνεργαζόμενα μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα ισχύσουν τα κριτήρια ε, του 1, που υπάρχουν στην διάταξη 1 παράγραφος 2 για τα δυτικά μέλη και αυτό θα καλυφθεί ε, και θα ισχύσει για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε συμβαστική πρόταση, θα την υποβάλουμε στην Ελληνική Προεδρία, ούτω ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα κατά αυτή την κοινοβουλική θετία ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Καρβάλια. Ε, κύριε Γιώχαντζεν ε, θέλετε να μιλήσετε κάτι, να πείτε κάτι εκ μέρους κάποιου σχεδόν συγκητού. Τι θέλετε, προσπαθείτε να ελκύσετε την προσοχή μου. Θέλω να λάβω το λόγο, αλλά όχι, δεν θα μιλήσω εκ μέρους κάποιου σκιώδους. Θέλω όμως το λόγο. Καλά, θα σας γράψουμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Έλλα. Σας ευχαριστώ. Θα ε, αναφερθώ σε δύο σημεία, σε δύο τμήματα. Καταρχάς σε ό,τι αφορά το δικαστικό. του Σε θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι αποτελεί ένα μεγαλύτερο πακέτο του πακέτο ε, επένδυση στην καινοτομία. Και είναι λοιπόν ένα τέτοιο πακέτο συναπόφαση. Τι σημαίνει λοιπόν στην παρούσα φάση. Η Ήτρε ψήφισε το πακέτο αυτό την προηγούμενο μήνα είχαμε αυτή την οριζόντια προσέγγιση και μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες περικοπές. Όχι επειδή θέλουμε να κάνουμε περικοπές, απλά να αποτυπωθούν και οι γενικότερες περικοπές του προϋπολογισμού του 5% που προτάθηκε από την ΙΤΡΕ. Ε, Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα οριζόντια αυτά θέματα, δείξαμε νομίζω πυγμή στο πρώτο τριμερή διάλογο και ε, δείξαμε ότι ε, ελέφθησαν υπόψη οι ανησυχίε του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο για τα θέματα συναπόφασης και ε, συμφωνής ε, διαβούλευσης μάλλον, έλεφθησαν υπόψη από, το, από την Επιτροπή. Το θέμα λοιπόν ήταν το χρονοδιάγραμμα. Ανεπίσημα έχουμε μία συμφωνία με την με το Συμβούλιο και την ε, Επιτροπή για να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία της πραγματεύση, στον τρομερή διάλογο. Γιατί αν παραμείνουν στο πακέτο διαβούλευσης, ναι. εμ, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα ληφθούν υπόψη σοβαρά από το Συμβουλίο, αλλά μας τελειώνει και ο χρόνος. Επί της ουσίας, ε, καταλαβαίνω ότι η συγκήτρια θέλει να ξανανοίξουμε το θέμα αυτό, γιατί γίνονται κάποιες έντονες προσπάθειες από τις ε, ισπανικές ε, εταιρείε να συγκαταλεχτούν και να χρηματοδοτηθούν. Δεν ε, υποθέτω ότι το θέμα είναι ουσία. Το θέμα είναι η αρχή. Αν το Κοινοβούλιο ξανανοίγει πακέτα τα οποία πέρασαν από διαπραγμάτευση μεταξύ Επιτροπής και της Βιομηχανίας πριν από τρία χρόνια, Τι θα γίνει δηλαδή με κάθε εταιρεία που τον υστέρων θα θέλει να συμπεριληφθεί σε έναν όμιλο εκ των υστέρων, θα μπορεί να το κάνει. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν με το 2, 15, 17 και 24 τις τροπολογίες αυτές, σε ό,τι αφορά δηλαδή να ανοίξει αυτός ο κατάλογος για τα μέλη χρηματοδότησης. Επίσης, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ισορροπία κατανομής. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια οριζόντια διάσταση η οποία προέρχεται από τους κανόνες, τον κανονισμό. Προσπαθούμε λοιπόν οι διαδικασίες για την εκχώρηση κονδυλίων να καταστεί πιο διαφανής. Και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν μένουν όλα αυτά στα ιδρυτικά μέλη μόνο και στη, στα χέρια της μεγάλης βιομηχανίας, της ισχυρής βιομηχανίας. Αλλά για να υπάρχει αυτή η ισορροπία, η συγγήτρια αυτό που προτείνει ουσιαστικά δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, την αλήθεια, όπως έχει διαμορφωθεί στο κράτο. Αυτό, αυτό στην πραγματικότητα. Αυτό θα σήμαινε ότι εκχωρούνται πιο πολλά κονδύλια σε τέτοιες επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι είναι σαφές λοιπόν ότι όλα τα τμήματα της, ε, του κλάδου και οι μικρομεσαίες καταλαβαίνουν ότι έχουμε την ε, ισορροπία αυτή σε αυτό 40% δηλαδή για τους, ε, τα ιδρυτικά μέλη, 30% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το καθεξής, ότι είναι ρεαλιστικό αυτό ως ε, κλίδα κατανομής. Αυτό λοιπόν έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές θα τα μπλέξουμε. Γιατί ουσιαστικά θα αναιρέσουμε αυτά που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια. Και είτε το Συμβούλιο δεν θα τα αποδεχτεί αυτά γιατί είναι φάκελος διαβούλευσης και κατά δεύτερον θα τίνεσαι και στον αέρα το χρονοδιάγραμμα γιατί κάθε επιτροπή θα πήγαινε και θα έκανε καταγγελία, θα έπρεπε να γίνουν διαπηρεσικές διαβουλεύσεις, δεν θα είμαστε έτοιμοι για την Ολομέλεια και τελικά θα καταλήξουμε στο δεύτερο κύμα και κατά πόσον ε, διατίθεται τέτοια κονδύλια το 2017 είναι κάτι το οποίο αμφισβητούμε ιδιαίτερω. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποτεχτούμε ότι έχουμε κάποιες οριζόντιες προτάσεις, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με προσοχή με τον εισηγητή και ρεαλιστικά θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στον τρέχοντα τριμμένη διάλογο. Ιδάλλως θα παραμείνει ένας φάκελος διαβούλευσης και δεν θα περάσει σε πραγματικό επίπεδο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Μιτάλ Κουαδράς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο τομέας των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι ανταγωνιστικός και πλευράς τεχνολογικής προχωρημένος, βρίσκεται σε φάση επέκτασης. Έχουμε επίσης κάποιες, διαγωνισμού ε, διαγωνισμούς που τους κέρδισαν διάφορα ευρωπαϊκά κονσόρτσια, όμιλοι επιχειρήσεων και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικής όπου οι επιδόσεις είναι επιδόσεις θρέμβου για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ισχύει πάντως εξίσου ότι υπάρχει άγριος νεονισμός από άλλες δυνάμεις και άρα δεν μπορούμε να επανεπαφθούμε στις δάφνες μας. Οπότε, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η κοινή πρωτοβουλία έρχεται την κατάλληλη στιγμή, εμείς θα πρέπει να την χαιρετήσουμε και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέβασε αυτή την πρόταση κανονισμού. Όπως είπε η συγγήτρια, θα πρέπει να βρούμε τι συνέργεια μπορεί να ισχύσει μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ούτω ώστε ο κλάδος των σιδηροδρόμων να είναι κλάδος εχμής, να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τους ανταγωνιστέ που προέρχονται από τον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή αυτής της έκθεσης Ο συγητής εργάστηκε με πίεση χρόνου, πάρα, πολύ καλά. Το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Για να δούμε τι βελτιώσει μπορεί να επιδέχεται, περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα ιδιωτικά μέλη. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι θα κάνουμε πριν τεθεί σε ισχύ να μην θεωρήσουμε ότι εδώ πέρα θα οδηγηθούμε σε διαμάχη και μονομαχία των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα, χρειάζεται όχι ανταγωνισμός, όχι κόντρα, αλλά κοινή προσπάθεια. Ακριβώς όπως προτείνει η εισηγήτρια και είναι πάρα πολύ εύστοχο. Και μας λέει ότι εδώ θα πρέπει να εμπλακούμε με το σύνολο του κλάδου και όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, άρα αυτό που λέει θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Να δούμε πώς θα έχουμε και επισεγγίσεις, ότι θα κατησχίσουν οι καλύτεροι, πιο άξιοι. Είναι επομένως πάρα πολύ φτωχή αυτή η πρωτοβουλία και πάρα πολύ χρήσιμη. Να στηρίξουμε επομένως το κείμενο της εισηγήτριας και να βιαστούμε ούτως ώστε πριν τις εκλογές να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδρομή της της έκθεσης. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και αυτή η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Καταρχάς, διότι υπάρχει προπτική επανεκβιομηχάνησης της Ευρώπης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία. Δεύτερον, από περιβαλλοντική σκοπιάς, πρόκειται για ένα βελτιστοποιημένο μέσο μεταφοράς ε, μικρών και μεσαίων αποστάσεων και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει σύγκληση όλων των κατασκευαστών σιδηροδρομικών υποδομών και όλων των χωρών για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα σε όλες τις γραμμές, σε όλες τις χώρες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες προκειμένου να εγκρίνουμε το ζήτημα αυτό στη διάρκεια της θητείας μας, διότι η βιομηχανική ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ευνοϊκές συνθήκες για να έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκούς διαχειριστές μεταφορών. Και έτσι να βελτιστοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές μεταφορές. Είναι σαφές ότι εμείς θα, θα είμαστε οι βασικοί χρήστες, διότι αν υπάρχει μια πραγματικά ευρωπαϊκή υπηρεσία υψηλής ταχύτητας, ελάχιστοι θα είχαν ε, ανάγκη να ταξιδεύουν με αεροπλάνο, θα ήταν ε, πιο γρήγορες οι μεταφορές και φυσικά λιγότερα. Ε, ενεργοβόρο από πλευράς χρήσης καυσίμων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, ταχύτατη έγκριση του συγκεκριμένου ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πιλάρ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι ε, πιέστηκε λόγω χρόνου κάτι το οποίο δεν συνέβη με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τις κοινέ επιχειρήσεις και επομένως ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτός ήταν ο μικρός αδελφός από χρονικής τουλάχιστον σκοπιάς που χρειάστηκε να γίνει πιεστικά και βιαστικά. Να σας πω ότι πράγματι πρόκειται για έναν από τους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη συνολική παρουσία Πολλές φορές αναφερόμαστε στην έλλειψη ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων ε, βιομηχανικών τομέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι εδώ αντιθέτως Πρόκειται για έναν ε, τομέα εχμής, ε, στον οποίο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει επανειλημμένως και αποδεικνύουν διεθνώς ότι έχουν μεγάλες δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και έχουν και διεθνή αναγνώριση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον τομέα αυτό. Σαφώς υπάρχει πίεση χρόνου, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ε, υπάρχει και πίεση ε, δυστυχώς για το shift to rail, αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει πίεση χρόνου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα, την δυνατότητα να ξεκινήσει ε, μια διαδικασία εδώ ώστε να αφήσουμε το σημάδι μας για μεγαλύτερη ε, συμμετοχή και διεύρυνση και άνοιγμα του τομέα αυτά σε αυτό τον τόσο ε, νευραλγικό τομέα. Γι' αυτό και εγώ από πλευρά μου θα υποστηρίξω οποιαδήποτε τροπολογία και πρωτοβουλία βελτιώσει το κείμενο. Ε, δεν γνωρίζω με πάσα λεπτομέρεια την πρόταση του κυρίου Οντή θα τη δω και νομίζω ότι μαζί με την πρόταση της εισηγήτριας και την πρόταση του κυρίου Οντή και με τις άλλες προτάσεις που ενδεχομένως θα λάβουμε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να συνδυάσουμε λίγο πιο αποτελεσματικά ε, τις προσπάθειές μου. Συμφωνώ και με τον κύριο Έλερ ότι θα πρέπει εμείς να χαράξουμε το δρόμο για να υπάρχει άνοιγμα για συμμετοχή και άλλων επιχειρήσεων. Very Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώχανσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποια σχόλια να κάνω καταρχά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το shift to rail, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να το δούμε ως μια ευκαιρία για να ενισχύσουμε την βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά είναι και ένα κομμάτι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές μας ανάπτυξη. Θα πρέπει να τονίσουμε και να ενισχύσουμε τη σύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης και μεταξύ του κόσμου στην Ευρώπη. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τις ε, απόψεις του κ. Έλερ σε ό,τι αφορά την επένδυση σε, άλλες, ε, σε άλλα τέτοια έργα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να φανεί ότι προαγάγουμε τέτοια το shift to rail παραπάνω από τα υπόλοιπα P2P ε, της πράξης δημοσίου-δημοσίου τομέα. Θα πρέπει λοιπόν όπου είναι αυτό δυνατόν να τηρήσουμε τις ε, οριζόντιες ε, διατάξεις που ισχύουν για όλο το πακέτο. Ιδάλλως πιο πολλά έχουμε να χάσουμε παρά να κερδίσουμε. είναι λοιπόν πιο συνολική η προσέγγιση μας. Σύμφωνο λοιπόν με αυτά που είπε ο κύριος Ήλερ. Και ασφαλώς έχει δουλέψει πολύ σκληρά σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές που άπτονται των άλλων πτυχών του πακέτου και θέλει λοιπόν όλα αυτά να έχουν μία συνοχή. Ξέρω λοιπόν ότι πολλά έχουν ήδη γίνει για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κάπως διστακτικός ό,τι αφορά την εισαγωγή νέων αλλαγών. Έχει συμφωνηθεί μια κατάσταση από την Επιτροπή και από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε βήματα προς το εμπρός, να προχωράμε, όχι να περιπλέκουμε υπερβολικά τη διαδικασία. Και το αναφέρομαι σε αυτά που είπε και ο κύριος Οντί που έδειξε κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι σκόπιμο να αλλάξουν οι προδιαγραφές για τις εταιρικές σχέσεις. Αυτό ενδεχομένως πιο πολλές δυσκολίες να προκαλέσει παρά να απλοποιήσει το οτιδήποτε. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω τώρα, σε ό,τι αφορά μία από τις τροπολογίες της εισηγήτριας, η υπαριθμό 16 συγκεκριμένα, η τροπολογία 16. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για ε, αμαξοστοιχείες υψηλής μεταφορικής ικανότητας. Εδώ όμως η ζυγήτρια μιλά για αμαξοστοιχείες υψηλής ταχύτητας. Υπάρχει μια διαφορά. Η υψηλή χωρητικότητα, η υψηλή ταχύτητα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Γιατί η συγκήτρια αναφέρει ότι αυτό θα συνάδει με τις υπόλοιπες ψηφοφορίες της ΙΤΡΑ για τα υπόλοιπα PPP. Γιατί λοιπόν να γίνει αυτό για το shift to rail. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των αμαξοστοιχείων υψηλή ταχύτητα και έχω κάνει πολύ lobbying αυτό στη Σουηδία. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα τρένα υψηλή χωρητικότητα είναι πιο αξιόπιστο και σε ό,τι αφορά τα φορτία. Δεν μα απασχολεί ιδιαίτερα, ξέρετε, τόσο πολύ πιο πολλά καλύπτονται με την υψηλή χωρητικότητα παρά με την υψηλή ταχύτητα. Να προσέξουμε λοιπόν με την ορολογία στο σημείο αυτό και επαναλαμβάνω ότι αυτό μα απασχολεί ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά και τι κοινωνικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σήμερα για τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και χωρών και κόσμου. Και αυτό επίση και σε ό,τι αφορά τον αγωνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώχανσον. Η κυρία Τράτμαν έχει Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais euh, euh, revenir sur θέλω να σχολιάσω τις οικονομικές συνθήκες να με το θέμα. Να και μετά από δύσκολες εννοήσεις για αυτό τον σημαντικό κλάδο καταλήξαμε εδώ σε αυτές τις συνθήκες της νέας όθησης των πραγμάτων και βέβαια είχαμε το Clean Sky και εκεί πρόκειψε κάποιο πρόβλημα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την ε, Ζωζέφα, τη συνάδελφο που επιτελεί σημαντικό έργο και συνεγέρασε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Πρώτα αυτά γνωρίζουμε ότι στο τσακ τα κατάφερε μετά από πιέσεις, από λόμπι, γιατί πρόκειται περί στρατηγική σημασία. Οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει όσον αφορά μια χρηματοδότηση μακρόπνοευδο ώστε να μπορέσουν οι εταιρείε του ιδιωτικού τομέα να έχουν εξασφαλίσει την οικονομική ισορροπία για να μπορέσουν να έχουν απόδοση επί τη βάση των επενδυσιών τους. Είμαι λίγο μπερδεμένη όσον αφορά κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτή, αυτό το σχέδιο κανονισμού και έχουμε αυτό το 40% των μελών που είναι 30% κάτι το οποίο σημαίνει ότι το 47,4% της, ε, της, ε, της Ευρώπης πάει στο 36 από το 47,4% οπότε αυτό είναι τώρα το θέμα το τι θα γίνουν οι επενδύσεις γιατί το συμφέρον των ε, πιο μικρών επιχειρήσεων που κινούνται στον κλάδο και χρειάζονται αυτή την πρωτοβουλία, δεν θα πρέπει ε, να, να αναφέρει διάσπαση του μετώπου το συμπίνο, οπότε θα πρέπει σε αυτή τη φάση να επιφυλαχθώ για το πόσο είναι στεγανή αυτή η πρόταση, γιατί δεν νομίζω ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να θέσει αμφιβόλο το οποίο έχει ε, συμφωνηθεί από αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία και ουσιαστικά δίνουμε ένα αντικίνητρο όσον αφορά την, ε, την αίσια κατάληξη αυτές τις διαδικασίες. Άρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν το βάρος των επενδύσεων θα μπορούν να το κάνουν αυτό ε, με όρους ε, που θα εγγυούν μια ισορροπία μεταξύ των δικών προσπαθειών και της Ευρώπης. Και έτσι να δούμε αν θα πετύχουμε. Οπότε άκουσα όλα αυτά τα θετικά για τα οποία συμφωνώ και θα πρέπει η ΜΜΕ που έχω και εγώ στην περιφερειά μου να μπορούν να σταθούν και για τα φόρτιγα τρένα αλλά και για τις αστικές περιοχές και ακριβώς θα πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τον κλάδο των φορτηγών τρένων να μπορούν οι επιχείρησει να κινηθούν σε μεγάλες γραμμές άρα θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο μεταξύ τους να μπορούν να συνεργαστούν προσοχή η απόφαση αυτή είναι στρατηγική σημασία και θα πρέπει να την λάβουμε με γνώμονα την εξασφάλιση των επιχειρήσεων. Um, is Πρόεδρος, θέλει άλλος συνάδελφος το λόγο, ο κύριος Σέλερ. Κυρία Τροσμάν, έχετε δίκιο. Πρέπει να βιαστούμε, αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί δεν είναι το θέμα απλώ το πώς θα ε, κατανοούμε τους πόρους με τρόπο σωστό μεταξύ ιδιωτικών μελών κλπ. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με την περικοπή των πόρων που έχουν διατεθεί. Αν πάρουμε μόνος από τα ιδρυτικά μέλη και από τους συνεργάτες ε, τους πόρους, τότε αλλάζει τελείως η ισορροπία της πρότασης. Ξοδεύουμε κυρίως δημόσιο χρήμα και όχι χρήμα των επιχειρήσεων. Οπότε τότε αναγκάζουμε τη βιομηχανία, το ξανασκεφτεί και θέτουμε εν κινδύνο ό,τι συμφωνήθηκε. Καταλαβαίνω ότι όλοι εδώ θεωρούμε ότι θα συμμετάσχει πλήρως και σε ευξημένο βαθμό η βιομηχανία και όχι το ανάποδο άσχετα από το ότι θα υπήρχε και το κοινωτικό χρήμα. Προσοχή εδώ, δεν πρόκειται για απλή ανακατανομή. Εδώ έχουμε περικοπή σημαντική της πρικοδότησης για την όλη πρόταση. Αυτά δεν προβλεπόντουσαν στην αρχή. Εμείς πιέσαμε ούτως ώστε να ε, στα δίστα πόδια της και πάλι αυτή η πρόταση, το shift to rail. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα θέτουμε να αμφιβόλο και εγκινδύνω τη δική μας πρόταση. Ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανείς άλλος. Ωραία, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπαρέα, για την έκθεση αυτή. Και να σας πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που καταβάλλατε για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και σκοπό έχει να συγκεντρώσει πιο μεγάλο ποσοστό του φορτίου και των επιβατών στους σιδηροδρόμους. Έχετε δίκιο, έχουμε ένα πακέτο για τους σιδηροδρόμους και θεωρούμε ότι το Shift to Rail είναι τεχνολογικός πυλώνας των προσπαθειών μας να δημιουργηθεί μια, ένας ενιαίος χώρος ευρωπαϊκός για τους σιδηροδρομούς. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να ενισχυθεί αυτός ο κλάδος και το ξέρετε αυτό. Αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε λοιπόν μια δέσμευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το συντομότερο δυνατόν θα τα εγκρίνουμε αυτά. Θα τα προωθήσουμε αυτά. Γιατί είναι μια σημαντική όθηση. Και σας παρακαλώ λοιπόν να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους σιδηροδρόμους και να τα περάσουμε αυτά γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, να πω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει την ε, συντριπτική πλειονότητα των ε, οριζόντιων τροπολογιών και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί σας. Μόνο μία κόκκινη γραμμή υπάρχει. Να σας την ανακοινώσω. Η τροπολογία υπερθμών 8. Και ο κύριος Οντή νομίζω είπε προηγουμένω ότι το shift to rail εγκρίθηκε μετά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και άρα είχε ήδη συμπεριληφθεί η περικοπή στην πρόταση και άρα άμα γίνουν επιπλέον περικοπές ουσιαστικά θα επιβαρυνθεί δύο φορές το shift to rail και μην την αποδεχτείτε λοιπόν αυτή την τροπολογία την υπερθμό 8 με τα υπόλοιπα δεν έχουμε τόσο θέμα, μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την τροπολογία 8, σας παρακαλώ, υποστηρίξτε μας και απορρίψτε την. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες τροπολογίες της κυρίας Μπαρία της Συγγητρίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Φυσικά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες τις οποίες δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Τα έχουμε εκθέσει, όπως είπε και ο κύριος Έλλη και η κυρία Τράουτμαν. Ε, ανέφεραν τα επιχειρήματα, δεν πρόκειται να τα επαναλάβω, αλλά να επαναλάβω ότι ήταν πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία την οποία διαπραγματευθήκαμε και την πετύχαμε μετά από πολλούς μήνες. Μην την θέσουμε ένα αμφιβόλο. 15, 17 και 24. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν δεν γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε όμως τις προτάσεις της και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση προτείνοντας νέο κείμενο στην τροπολογία 19 όπου επί της αρχής δεν αποδεχόμαστε τις τροπολογίες της ηγήτριας σε ό,τι αφορά τις εξουσίες προς το ΕΡΑ. Καταλαβαίνουμε όμως το σημείο στο ΣΥ που αναφέρει ότι τα μέλη τα οποία πληρούν ως ε, μοναδική ε, νομική οντότητα, τα κριτήρια που αναφέρονται στο 1-2 θα εκπροσωπούνται αυτόματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο εδώ. Και αυτό είμαστε επιτευχμένοι να το διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο προκειμένου τα μέλη, τα συνεταιριζόμενα να έρθουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα ιδρυτικά μέλη να συμμετέχουν στο ίδιο βαθμό και να εκπροσωπούνται αυτόματα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ω εκ τούτου πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει μία λύση. Και αυτό και προτείνουμε προκειμένου να επιλύσουμε το θέμα αυτό με την τροπολογία που προτείνει η συγκεκριά. Δεσμεύομαι λοιπόν αυτό και σας το αναφέρω. Συμφωνώ με τον κύριο Έλετον, τον κύριο Ντίκ, την κυρία Τράουτμαντ να επαναλάβω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η περικοπή από πλευρά του προπολογισμού και η αναλογία 40-30% το άνοιγμα του, της κλειστής λίστας στο παράδειγμα 1 δεν είναι αποδεκτό, αλλά όλες οι υπόλοιπες ε, προτάσεις προκειμένου να δοθεί μια ενίσχυση στον συνδρομικό κλάδο μας βρίσκουν σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η συγγήτρια για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τα ενθαρρυντικά τους λόγια, ε, για την πίεση χρόνου που είχαμε για την ε, παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Είναι αλήθεια ότι δεν μας δόθηκε πολύς χρόνος, χρειάστηκε να τρέξουμε πολύ και προσπαθήσαμε παρόλα αυτά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και το λέω αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταλάβει ότι και εμείς χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε το ζήτημα. Ας τα δούμε λίγα-λίγα τα θέματα. Ο κύριος Σοντή, μέσω της κυρίας Καρφάλιο, μας είπε την άποψή του. Η έκθεση αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης δέσμης ε, εκθέσεων και ε, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες οι οποίοι έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων και δεν μπορούμε εμείς να τους αλλάξουμε εδώ και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζει η πλειονότητα των πολιτικών ομάδων. Δεν μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να ξανασυζητάμε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να καθυστερήσουν και εν μέρει όλες τις ε, σχετικές πρωτοβουλίες και κυρίως μια τέτοια πρωτοβουλία. Αναφερθήκαμε στη σημασία τη έγκαιρης έγκρισης αυτής της έκθεσης, στη διάρκεια αυτής της θητείας. Συμφωνώ απολύτως. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μακρηγορήσουμε και να χάσουμε και άλλο χρόνο. Αυτή τη στιγμή ε, ε, υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης και διαφάνειας. Και επίσης ε, καταρχάς θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο θέμα της υψηλής ταχύτητας και υψηλής χωρητικότητας. Ίσως έπρεπε να το αναφέρουμε, δεν ξέρω ίσως που εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε και την υψηλή ταχύτητα που δεν αναφέρεται εδώ πέρα ως κάτι πολύ σημαντικό θα το ξαναδιαβάσω και θα, διαβάσω, θα απαντήσω απευθεία ε, στον ε, συνάδελφο που το σχολίασε, αλλά εμείς θα θέλαμε να αναφέρεται και η υψηλή ταχύτητα στην έκθεση αυτή. Και θα ήθελα τώρα να σταθώ στα δύο θέματα που από ό,τι φαίνεται ανησυχούν ε, τους συναδέλφους και ανησυχούν μέχρι του σημείου να πείτε ότι το έχω κάνει εκ εγώ ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να συμμετέχει η τάδε η δίνα επιχείρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έδωσα απλώ έναν ενδεικτικό κατάλογο και μου φαίνεται απίστευτο να υπάρχει ένα κλειστό κατάλογο πριν υπάρξει συνένεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την έκθεση αυτή. Θεωρούμε και το λέω σαφέστατο, ε, όπως είπε και ο κύριος Έλερ, ότι τα θέματα τα οποία έχουν ήδη αποφασιστεί από την Σύμπραξη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι θέματα τα οποία δεν μπορεί να συζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αρχή διαφάνειας και να υπάρχουν δυνατότητες για άλλες ευκαιρίες και θεωρούμε ότι αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι ενδεκτικός και όχι πλήρης. Και το θέμα που έθεσε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονός ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση ασαφή το ιδρυτικό μέλος και ε, τα συνδεδεμένα μέλη. Ε, πώς θα συσχετιστούν αυτοί οι δύο, τι δικαιώματα θα έχουν τα συνδεδεμένα μέλη. Όλα τα συνδεδεσμένα μέλη θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κλητήρια. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι ο κατάλογος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αυτό ως το οποίο θα καθορίσει τις στρατηγικές γραμμές και το ε, διευθυντικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι κλειστός κατάλογος. Όταν ε, ε, ε κλείσει, όταν εγκριθεί η έκθεση θα πρέπει να πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άποψη και πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν είναι δυνατόν να είναι προαποφασισμένο. Κάτι πρέπει να πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα ε, μας είπε ο κύριος Έλερ ότι είναι προαποφασισμένο. Δεν γίνεται. Πρέπει και εμείς να αποφανθούμε. και τι γίνεται για τη συμμετοχή. Ζητάμε 10% από τα ιδρυτικά μέλη, το συζητήσαμε και αυτή τη στιγμή το να υπάρχει ένας κλειστός κατάλογος ε, για, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδρυτικών μελών και ένα 10% για να το δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτούς τους ανθρώπους που λέμε ότι πρέπει να συμμετέχουν και ότι είναι το μέλλον της Ευρώπης. Τα λέμε συνεχώς. 10% η ισορροπία είναι το ίδιο. Φτάνουμε στο 100%. Απλώς κάναμε ένα καταναμή. Δεν τροποποίησαμε τίποτα και πραγματικά εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο η κατάσταση να συγκρατηθεί κάπως, δεν χρειάζεται αντιπαράθεση, ο διάλογος αρκεί, και πρώτον αυτό, και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει δώσει ένα κλειστό κατάλογο, το είπαν εδώ και κάποια μέλη, και τώρα προσπαθεί να μας δώσει μια εναλλακτική λύση που είναι ένα... Μια σαφής κατάσταση, είναι σε λίμπο. Έχουμε κάποια συνδεδεμένα μέλη τα οποία δεν θα έχουν ε, ιδέα τι ακριβώς ε, δικαιώματα και υποχρεώσεις θα έχουν. Και ε, ο σιδηροδρομικό τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι μεταφορέ τη Ευρώπη και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το σκεφτεί και θα πρέπει να λάβει υπόψη και ότι πρέπει να έχει άποψη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να συνενέσει σε οτιδήποτε αποφασίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τώρα θα ήθελα να πω το εξή. Νόμιζα ότι τα πηγαίνουμε καλά και ότι τηρούμε το χρονοδιάγραμμα όπως και πρέπει φυσικά σε τέτοιε συζητήσει, αλλά θα ήθελα να κάνει μια περαιτέρω παρέμβαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη δίνω λοιπόν το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα απλά να διευκρινίσει δύο στοιχεία μετά από την παρέμβαση τη συγγήτρια. Το shift to rail και ο κλειστό κατάλογο, η κλειστή λίστα δεν ήταν ιδέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 19 που απορρίζεται ότι χρειαζόμαστε αρκετές, αρκετούς πόρους και ιδιωτικούς και δημόσιους για την πρόταση τέτοιων πρωτοβουλειών. Αυτό λοιπόν να το διευκρινίσουμε. Από το άρθρο 19 του ορίζοντα 2020 σε ό,τι αφορά τα συνδεδεμένα μέλη και τα δικαιώματά τους, όπως είπα και προηγουμένως και παρέθεσα ότι τα συνδεδεμένα μέλη ως νομικές οντότητες αυτόματα θα συμπεριλαμβάνονται, στο, θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον δηλαδή έχουμε καταθέσει τα ίδια χρήματα. Δεν είναι κλειστό λοιπόν σε αυτά τα μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης να πω ότι σε ό,τι αφορά τα τρένα υψηλής ταχύτητας συμφωνεί μαζί σας η, και η Επιτροπή, η κυρία να συμπεριληφθεί και αυτά. Αλλά θέλουμε και τα περιφερειακά τρένα. Άρα στην 16 προτείνουμε να αναφέρεται ή και τα τρένα υψηλή ταχύτητα. Και σε ό,τι αφορά τι οριζόντιε περικοπέ, πιστεύουμε ότι το shift to rail ασφαλώ περιλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα τη πρωτοβουλία, αλλά δεν χρειάζεται να συμμετέχουν ένα τμήμα όλων των, του πακέτου και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρυνθούν διπλά από τις περίκοπες. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την καινοτομία στον κλάδο αυτό που είναι πολύ απαραίτητη προκειμένου να... Και θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να ξεπεράσει κάπως τα εμπόδια προκειμένου να προχωρήσει με ταχύτητα αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Να σας πω ότι από το σύνολο των επιχειρήσεων μόνο μια επιχείρηση έχει κλειστό κατάλογο σαν αυτό που έχουμε στο Shifty Rail. Ε, δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας, αλλά θα ήθελα να δω και ένα κείμενο ε, υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμμετέχουν αυτά τα συνδεδεμένα μέλη και ποια κριτήρια των ιδρυτικών μιλών πρέπει να πληρώνουν. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση για την έκθεση αυτή και θα ήθελα για να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα 5η 20 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για να μπορέσουμε να ε, ψηφίσουμε στις 18 Μαρτίου στην Επιτροπή και να περάσει η έκθεση από την Ολομέλεια του Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτουμε για δύο λεπτά και θα ψηφίσουμε στις 10 ακριβώς. Okay, the committee will come to order. Ξαναρχίζουμε την συνεδρίαση και πάμε στο επόμενο θέμα μας διατάξεις που είναι οι ψηφοφορίες. Όλοι, παρακαλώ, να βγάλετε την κάρτα της ψηφοφορίας, να την τοποθετήσετε στην συσκευή και θα κάνουμε πρώτα-πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. προτείνετε. Να κάνουμε να μην κάνουμε διάλειμμα για καφέ. Ψηφίστε ναι ή όχι. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι. That's number of cards. Yes. That's, sorry, that's, that's, okay. All right. Vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας. Α, εσείς συνάδελφοι δεν έχετε την κάρτα, οπότε θα λάβουμε υπόψη του τι έχετε να ψηφίσετε κατά όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο πρώτο προσψήφιση θέμα που είναι το πρόγραμμα υποστήριξης για επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος. Η συγγήτρια είναι η κυρία Άντερς Ντότερ. Είναι διαδικαστικό. Δεν έχετε την ε, κάρτα σας. Τι θέλετε, αν θέλετε το λόγο μετά. Όπως ε, μπορεί να διευθυνθεί, δεν είμαι κυρία Αντεστότερα, αλλά για λογαριασμό τη, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή και το Συμβούλιο, γιατί ήταν μια άριστη συνεργασία μαζί της για την εκθέση αυτή. Οπότε και πάλι ευχαριστή κυρία Άντερ Ποιοι είναι υπέρ, λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, γι' αυτό και είπα για τις κάρτες. Και ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 32-1. Συν άλλες δύο ψήφοι υπέρ, άρα 34 υπέρ. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια προς την κυρία Άντες Ντότερ. Τώρα, επέκταση της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Κοινότητας Ένωσης Τελοσμάνων και Ενωμένων Πολιτειών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 27 υπέρ. Συν 2. Α, εσείς έχετε και ψηφίσατε. Ωραία. Τότε 28 υπέρ, 2 κατά και 4 εποχές. κρίνεται επομένως. Σας ευχαριστώ. Και εδώ ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες. Μπορεί να φύγει όποιο θέλει να πάει, να προλάβει το τρένο ή το αεροπλάνο, οτιδήποτε. Α, τι έχετε εσείς, διαδικαστικό. Πρόεδρε, λέει ο κύριος. Έλα. Να πρέπει να βάλουμε σε κάποια μέρη σε διάταξη, να ανταλλάξουμε απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την επερχόμενη συμφωνία με την Ελβετία ε, Πρόεδρο. Ναι, αλλά ποιος θα μπορέσει να πάει στην Ελβετία για να δεχτούν για να το συζητήσει. Πάμε παρακάτω. We now come to, or I'll, you're all leaving very quietly, so we'll, we'll press on. Uh, we now come to the um, τροποποίηση της οδηγίας για συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίες για μείωση κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών. Ο κύριος Μπερτότ δεν μπόρεσε να παραστεί, αλλά ανταυτού θα λάβει το λόγο που αδειμονεί η κυρία Ιόντον. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας διαβάσω τι πρεσβεύει ο εισηγητής μας. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτό που διαβάσω. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, σεβαστείτε τον ε, εισηγητή και αν θέλετε κάτι να κουβεντιάσετε, παρακαλώ να το πράξετε εκτός της αιθούσης. Ή να συζητήσετε σιγά και να μην ακούγεστε. Όλα αυτά σας τα λέω από πλευρά του κυρίου Μπέρτο που είναι συγητής. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τροποποιήσει την ε, πρόταση όσον αφορά σκευασίε και προϊόντα συσκευασία για τη μείωση των αδρασίλων των πλαστικών σε Και οπότε θέλουμε εδώ πέρα να στοχεύσουμε στα προϊόντα τα οποία είναι μεταξύ 11 και 15 μικρών. Και αυτό νομίζουμε ότι είναι ο πιο κοινό τύπο σακούλα μεταφορά. Για να μπορέσετε να έχετε μια ιδέα για το φαινόμενο, θα πρέπει να σα πω για κάποιο, υπάρχουν κάποια στοιχεία του 2010 το ότι κάθε ε, Ευρωπαίο χρησιμοποιεί και πετάει κάθε χρόνο 198 πλαστικές σακούλες. 90% είναι λιγότερο σε πάχος από 15 μικρών. Και έχει αυξηθεί η χρήση και, και λόγω της διάδοσης πάνω των 10 δισεκατομμυρίων τέτοιων ε, σακουλών που και αυτό έχει συνέπειες σημαντικές για το περιβάλλον και για τις θάλασσες Ευρώπης. Ο βασικός στόχος που θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την οδηγία είναι να δούμε πώς θα μειώσουμε αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της κατανάλωσης και της χρήσης αυτών των σακουλών και να είναι οι χρήστες πιο υπεύθυνοι και να μην έχουμε επίσης απόρριψη τέτοιων ε, ε, σακουλών και να έχουμε καλύτερη χρήση των πόρων και οι πιο σημαντικές τροπολογίες που έχει αυτή η οδηγία έχει τα ε, βιολογικά προϊόντα και εκεί που χρησιμοποιούν το στοιχείο 134-32. Το, το πρότυπο 134-32. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθεί η βιομηχανία προς μια ανάκαμψη και θα στηρίξουμε τις προτάσεις, τις προσπάθειες των μελών, τόσο ώστε να ξανααποκτήσουν ως βιομηχανία ανταγωνιστικότητα. Μέχρι το 2020 ο όγκος το τέτοιων ε, χημικών ε, προϊόντων όπως και διαλυτικά και διάφορες χημικές ουσίες πρόκειται να ανέβει στο 7,3%. Αυτό θα είναι ε, κάτι που θα σημαίνει επιπλέον έσοδα 40 δις ευρώ και αυτό σημαίνει 90.000 θέσεις και αντίστοιχες ευμενείς συνέπειες έμεσες και θέλουμε μέσα σε δύο χρόνια από τότε που θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία να έχουμε τη χρήση σακουλών από 11 μικρών έως 19 γιατί και σακούλες των σούπερ μάρκετ επίσης να καλύψουμε και θέλουμε πάρα πολύ ε, λεπτές σακούλες επίσης να θέσουμε σε εμπορία από 1 έως 10, τι λέει εδώ πέρα, δεν ξέρω λέει μάλλον εννοεί και αυτό να χρησιμοποιείται και για τα φρούτα και λαχανικά στα σούπερ μάρκετ. Και εδώ πέρα λέει ο εισηγητή ότι θα τεθούν σε χρήση αυτά τα μέτρα επιτρέποντας στον κλάδο να βρει εναλλακτικές. Υπάρχουν αυτά τα πρότυπα και να μην έχουμε υπορβολική χρήση συσκευασιών. Οπότε να μπορέσει ο κλάδος να έχει χρόνο, να βρει εναλλακτικές λύσεις, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα τρόφιμα να μην υφίστανται περιβολική συσκευασία, αλλά να τηρούνται οι διατάξεις που στατεύουν την υγεία και όσον αφορά αυτές τις ελαφρές σακούλες μεταφοράς, Θέλουμε να τις αντικαταστήσουμε τελείως. Με ανακυκλώσιμο χαρτί και με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ελαφρές σακούλες. Να χρησιμοποιούν για κρέας, νοπό, ψάρια και αυτά τα είδη να εξαιρούνται από αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει ισχύσει το πρότυπο 13432 του 2002 και αυτές οι σακούλες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι για κάποιους βιολογικά απόβλητα σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. Όλα αυτά τα μέτρα της ε, οδηγίας θεσπίζουν κάποιους νέους κανόνες για καταναλωτές, σούπερ μάρκετ, ομοιογενός και έτσι να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. This was the, the opinion of, um... Και αυτή ήταν η γνώμη του εισηγητού μας, του κύριου Μπερτότου. Thank you very much uh, for that. Ευχαριστούμε πολύ. I now turn to Mr. Prodi. Και τώρα να δώσω το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αναφέρω λίγο τις αρχές βάσει των οποίων υπέβαλα τις τροπολογίες μου. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιους ορισμούς. Bio-based σημαίνει ότι η πρώτη ύλη είναι βιολογική, είναι βιομάζα, αλλά αυτό δεν αποτελεί απαραίτητο εγγύηση ότι το προϊόν θα είναι βιοδιασπόμενο και θα υπάρχει δυνατότητα κομποστοποίησης. Αυτές είναι ιδιότητες οι οποίες καθορίστηκαν από το ευρωπαϊκό πρότυπο και επομένως αποτελούν και τη βάση μιας πρότασης που θα πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι αυτές οι τόσο ελαφριές σακούλες έχουν μια πάρα πολύ σημαντική λειτουργία, διότι εγγυώνται προστασία από ε, απορρίμματα, από τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν ίσως να ε, βγουν από τη σακούλα και επομένως μας επιτρέπουν ε, να έχουμε καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να την κάνω αυτή την επισήμανση λοιπόν για το πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι σακούλες διότι Διαφωνώ. Στην αδιάκριτη φορολόγηση όλων αυτών των ε, συσκευασιών στον ε, ε, χώρο καταγωγής. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε συνολικά σε πλήρη βιοδιασποσιμότητα και δυνατότητα ε, βιολογικής κομποστοποίησης. Αυτό είναι που προέχει, διότι Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί δεν θα πρέπει να ε, επιβάλλουμε φραγμούς ε, στην εμπορική τους χρήση. Το σημαντικό είναι να υπάρχει πλήρης εξαφάνιση όλων αυτών των συσκευασιών που δεν είναι βιοδιασπόμενες και δεν υπάρχει δυνατότητα βιολογικής κομποστοποίησης και να χρησιμοποιούμε πλέον υλικά τα οποία μας προσφέρουν αφενών σε αυτή τη βεβαιότητα ότι υπάρχει προστασία και αφετέρου είναι και περιβαλλοντικά βιαδιασπόμενες. Επομένω, θέλουμε σακούλες που δεν σπάνε και δεν ανοίγουν και που είναι βιοδιασπόμενες. Αυτό είναι που έχει σημασία και αυτές οι βιοδιασπόμενες σακούλες επειδή ακριβώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και για ε, πιο υγρές τροφές, μπορούν να βελτιώσουν και τη συλλογή των ε, πιο υγρών τροφίμων, τα οποία εξορισμού είναι βιοδιασπόμενα. Υπάρχει λοιπόν μία συνέπεια και μπορούν να διευκολύνουν και τη συλλογή των απορριμμάτων. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε σακούλες οι οποίες ε, είναι συμβατές και μάλιστα βελτιώνουν και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και ότι στη συνέχεια θα διασπαστούν πλήρως. Υπάρχουν λοιπόν ήδη τέτοιες σακούλες οι οποίες είναι στη διαδικασία της έγκρισης και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεκτικό και βιώσιμο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάση. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, να ευχαριστήσω και την κυρία Τζόρνταν. Πού εκπροσωπεί τον εισηγητή σήμερα εδώ. Να τους ευχαριστήσω λοιπόν για τη δουλειά που έχουν κάνει. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κάποιο τρόπο είναι ευπρόσδεκτη. Αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά στεναρή. Και δυστυχώ πρέπει να πω ότι και ο εισηγητής της Επιτροπής Βιομηχανίας και η πρότασή του, το σχέδιο του κειμένου του θεωρώ ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετά στεναρός. Για το πρόβλημα αν γέννη. Η κυρία Τζόζαν αναφέρθηκε ήδη στον τεράστιο αριθμό πλαστικών σακούλων που μολύνουν το περιβάλλον. Να προσθέσω στο σημείο αυτό ότι στη Βόρεια Θάλασσα έχουν γίνει μελέτες για τα θαλάσσια πτηνά και αν του 90% των θαλάσσιων πτηνών και των γλάρων έχουν λοιπόν στο πεπτικό του σύστημα ε, πλαστικές σακούλες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπολογιστεί ότι αναμίλη μπορεί να βρει κανείς ε, και ξεβράζουν στην ε, ακροθαλασσιά 72 σακούλες αναμίλη. Τα κομμάτια αυτά πλαστικού είναι εξαπλάσια από το πλανκτόν στην επιφάνεια της θάλασσας. Μιλάμε για ένα τεράστιο λοιπόν ε, περιβαλλοντικό πρόβλημα και θα πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ, όπως σας είπα, ότι είναι υπερβολικά ε, αδύναμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλά νομικά υποστηρίζει τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία θέλουν να πάρουν μέτρα εθνικά. Δεν ενθαρρύνει με κανέναν άλλο τρόπο. ούτε δίνει κίνητρα για την ε, ε, κατάργηση της πλαστικής σακούλας. Συμφωνώ και με την κυρία Άουκεν. Σε ό,τι αφορά τους δεσμευτικούς στόχους. ακριβείς ε, στόχους σε ό,τι αφορά και την τρέχουσα κατανάλωσή τους της πλαστικής σακούλας. Σε χώρες λοιπόν όπου είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση της πλαστικής σακούλας, ο στόχος είναι πιο υψηλός και αντιστρόφος. Αυτό μας φαίνεται ότι είναι, ίσως να φαίνεται μάλλον σκληρό, αλλά σε όλες τις χώρες που έχει δοκιμαστεί το σύστημα, Όταν επιβάλλεται μια τιμή για την πλαστική σακούλα, ο περιορισμός της χρήσης της πλαστικής σακούλας ήταν πραγματικά πολύ σημαντικός. Κάποια πιο λεπτομερή σχόλια, λοιπόν, για τις τις σακούλες, τις ελαφριές ε, σακούλες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για οργανικά απόβλητα. Η τελευταία ε, τροπολογία που προτάθηκε από τον εισηγητή της ΙΤΡΕ. Συμφωνώ να γίνει διάκριση μεταξύ της παραδοσιακής ε, πλαστικής σακούλας, αν μου επιτρέπετε τέλος πάντων αυτός ο όρος, και του μη οργανικού πλαστικού και των πραγματικά βιοδιασπόμενων πλαστικών. Νομίζω όμως ότι η διάκριση που προτείνει ο εισηγητής δεν είναι επαρκώς σαφής. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και τα οξοδιασπόμενα πλαστικά. Είναι ένα είδος βιοδιασπόμενων. it doesn't, uh, διασπάται σε πιο μικρά κομμάτια, τα οποία δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι, αλλά τα οποία επίσης είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Είναι εξίσου επιβλαβή για το περιβάλλον και για τα ζώα. Και συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Άουκεν, την εισηγήτρια από το, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι τα οξοβιοδιασπόμενα θα πρέπει και αυτά να καταργηθούν και να απαγορευτούν τελείως και να πρέπει να αντικαταστηθεί με τον Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο είναι ο κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ εκπροσωπώ τον κύριο Κρόιτσμαν, ο οποίος ε, είναι ο από την ομάδα μα για την έκθεση αυτή και δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα σήμερα και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω και να πω δύο λόγια εκ μέρου του. Καλώς ορίζω την πολύ ισορροπημένη ε, γνωμοδότηση του εισηγητή σε απάντηση Προ την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Θα ήθελα να κάνω κάποιε μικρέ παρατηρήσει όμω και πιστεύω ότι η συζήτηση για την πλαστική σακούλα θα πρέπει να ξεκινάει από την αρχή ότι υπάρχει πραγματικά όφελος από το να μειωθεί το πλαστικό και τα απόβλητα πλαστικού, αλλά από την άλλη να μην μπούμε και σε μια διαδικασία να τα κατηγορούμε για όλα, γιατί υπάρχουν και πλέον εκτήματα. ανάλογα με τις χρήσεις, πρέπει να αναρωτηθούμε και ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Ίσως αυτό θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ναι. Ε, ήμασταν σε έναν κόσμο που θα χρησιμοποιούνταν λιγότερο η πλαστική η σακούλα. Τι θα χρησιμοποιούσε ο καταναλωτής. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ερευνήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι θα γινόταν στην περίπτωση αυτή και ποια θα ήταν και ποιο θα ήταν τελικά ο συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μήπως θα χρησιμοποιούσαμε λιγότερο πλαστικό, αλλά θα κόβαμε πιο πολλά δέντρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας ανησυχεί κάπως και από πλευρά της Επιτροπής Περιβάλλοντος το ακούσαμε. Μπορεί να πούμε ότι στα πλαίσια της δικουρικότητας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιορίσουν την κατανάλωση της πλαστικής σακούλας. Ε, εδώ και χρόνια όμως βλέπω μια λυπηρή τάση σε ό,τι αφορά την ιστορική αγορά και σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα μεταξύ των κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι πρέπει αυτός να είναι ο σκοπό μας, γιατί σε τελική ανάλυση τελικά θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση κατακαιρματισμένη. Στην μία χώρα θα απαγορεύονται οι σακούλες, στην άλλη χώρα θα επιτρέπονται. Αυτό εξυπηρετεί το περιβάλλον επόμενο επιχείρημα που ήθελα να αναφέρω. Σίγουρα δεν είναι καθήκον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει ε, μια τιμή για την πλαστική σακούλα. Και τέλος, θα πρέπει να ελέγξουμε στη συζήτηση αυτή να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τα απόβλητα και μιλάμε για ένα προϊόν, την πλαστική σακούλα. Υπάρχουν λοιπόν προδιαγραφές ανακύκλωσης, υπάρχουν σχετικές οδηγίες οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς και ίσως λοιπόν καλύτερα θα ήταν να φροντίσουμε η νομοθεσία για τα απόβλητα και τα απορρίμματα να εφαρμοστεί εξίσου σε όλα τα κρατημέλη, προτού αρχίσουμε και συζητάμε μεμονωμένα προϊόντα. Ενδεχομένω λοιπόν να πετύχουμε καλύτερα το στόχο μα με τον τρόπο αυτό από το να ξεκινήσουμε να νομοθετούμε για μεμονωμένα προϊόντα. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Φανέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά έχουμε ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προοδεύσει, να προοδεύσει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, να προοδεύσει σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων συμφεράντων, σε θέματα προστασίας της ζωής των ζώων, σε θέματα προστασίας της βιομηχανίας και της έρευνας. Και εμείς αντί να προχωρήσουμε ε, σταματάμε γιατί δεν ξέρουμε αν θέλουμε να, πάμε, να μείνουμε στο μπροστινό πανδοχείο ή στο, πίσω πανδοχείο. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε μάχη για να φτιάξουμε χάρτινες σακούλες. Στην Ευρώπη υπάρχουν πλαστικές σακούλες πλήρως βιοδιασπούμενος που φτιάχνονται από το φλοιό της πατάτας ή του, από αραβοσίτη. Επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε την έρευνα, τη γεωργία και τη βιομηχανία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Γιατί αυτό το οποίο δεν λέμε εδώ στην Επιτροπή μας είναι ότι ήδη οι προτάσεις δεν αρκούν διότι έχουμε την αίσθηση ότι απλώς υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της πετρελαϊκής βιομηχανίας στην Ευρώπη διοργανώνεται ουσιαστικά η σπάνιδα πρώτων υλών. Πρώτων υλών για την κατασκευή ε, πλαστικής σακούλας θα οργανώσουμε με την κατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες ε, ε, φτιάχνουν πλαστικές σακούλες σε ε, χώρες στις οποίες υπάρχει χαμηλότερη μισθός για το εργατινομικό δυναμικό, φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Προσπαθούμε λοιπόν να επιβάλλουμε σακούλες που είναι επικίνδυνες για τα ζώα και για τους ανθρώπους. Η φοροαπαλλαγή για πλήρως βιοδεσπόμενες σακούλες, οι οποίες συνάδουν πλήρως και μπορούν να συνδυάσουν βιομηχανία, γεωργία και ε, προστασία του περιβάλλοντος, είναι η κατάλληλη λύση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να προσπαθούμε ε, να αλλάξουμε τα πράγματα. Αν ο καθένας θέλει να αγοράζει αυτό που θέλει, ναι, να το κάνει. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός αλλά ο ανταγωνισμός για τα πετρολαϊκά προϊόντα θεμελιώνεται στο γεγονός ότι εμείς ουσιαστικά οργανώνουμε την έλλειψη πρώτων υλών για να επιβάλλουμε συγκεκριμένους τιμούς, τιμές. Διαδιασπόμενες ακούλες μας επιτρέπουν να έχουμε προσέγγιση της γεωργίας και της βιομηχανίας και θα κάνουμε και κάτι καλό για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέρκη τώρα. Με τα χαρά σας δίνω το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Συζητούμε συμβιβαστικέ τροπολογίε για την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για το θέμα ακριβώς ε, που συζητούμε. Οι πλαστικές σακούλες δεν είναι τόσο θέμα απορριμμάτων και ούτε θέμα αποδοτική χρήση των πόρων. Είναι θέμα Απορριμμάτων, λέει ο Μιλήτρια. Πολλές φορές ε, μπορεί να επηρεάζουμε ε, πολιτικά μέτρα, ε, όχι πάντα. Βλέπουμε κάποιες πρωτοπόρες χώρες όπως η Φιλανδία και η Ιρλανδία οι οποίες χρησιμοποιούν 300 φορές λιγότερες σακούλες από άλλες χώρες και αυτό μάλλον οφείλεται σε τα κατάλληλα πολιτικά μέτρα. Συμφωνώ με το συντάκτη της γνωμοδότησης για την απαγόρευση των ελαφρών ε, συσκευασιών, αλλά γίνεται και μία συζήτηση για απαγόρευση το 2019 το 2020 και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δεχθούμε απαγόρευση για όλες τις μη βιοδιασπόμενες σακούλες κάτω των 2.000 χιλιοστών και επίσης ε, για ε, όλες τις βιοδιασπόμενες κάτω των 50 μικρών στο σημείο πώλησης. Υπάρχουν συνέπειες και για τη θάλασσα, για τις παρακτές περιοχές και για τον τουρισμό φυσικά. Και το θέμα είναι ότι αυτές οι πολύ λεπτές σακούλες δεν περιλαμβάνονται την παρούσα έκθεση. Γίνεται συζήτηση για εξαίρεσή τους. Ε, είμαι ανοιχτή σε συζήτηση, αλλά προς το παρόν θα ήθελα να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στόχο το 80%. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πολύ λεπτές σακούλες ε, και η ίδια η οδηγία για τις συσκευασίες έχει ε, άμεση υποχρέωση και συμφωνώ και με κάποια άλλα σχόλια τα οποία έγιναν, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει αυτή η νομοθεσία ε, να εξεταστεί ξεχωριστά από το όλο θέμα των απορριμμάτων, διότι ε, θέλουμε να εφαρμοστεί με σωστό τρόπο η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ε, και αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων βλέπουμε ότι κάποιες παλιές ιδέες ε, μεταφέρονται στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις σακούλες και η νοοτροπία μας θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και κάποιες ε, πιο καινοτόμες ιδέες. Κάποιος πρότεινε να χρησιμοποιούμε δίχτυα αντί για σακούλες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολες ε, ίσως στη διάσπασή τους και φυσικά απαιτούν και λιγότερο υλικό. Βλέπουμε επίσης ότι πολλές σακούλες χρησιμοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και των λιανικών πωλήσεων και ο πρώτος μας στόχος θα πρέπει να είναι να ε, στοχεύσουμε όντως στον τομέα των λιανικών τροφίμων και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται με τους άλλου κλέδου. Ε, για παράδειγμα, στις διαδικτυακές πωλήσει χρησιμοποιούνται πλέον ε, κατά κόρον πλαστικές σακούλες, οι οποίε είναι πολύ πιο χοντρές και ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο επόμενο στάδιο. Μετά από το 2020 λοιπόν για τα ε, λιανικά τρόφιμα. Τώρα, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται για τις μη βιομηχανικές συνθήκες. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί ορισμοί για τις βιοδιασπόμενες σακούλες και το θέμα είναι ότι δεν είναι όλες ε, διασπόμενες, διότι κάποια τμήματα θα παραμείνουν. Αν πραγματικά επιθυμούμε βιοδιασπόμενες σακούλες, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος ορισμός. Υπάρχει, για παράδειγμα, η οξοβιοδιασπόμενη σακούλα, η οποία δεν είναι ακριβώς βιοδιασπόμενη και δεν είναι πλήρως βιοδιασπόμενη και θα πρέπει ε, βαθμιδών να εξαφανιστούν αυτές οι σακούλες, ε, όπως ε, είπε και ο συνάδελφος Πρόντι. Έγινε και ολόκληρη συζήτηση για το θέμα της επικουρικότητας. Είναι πολύ καλή η συζήτηση αυτή, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση σε πλαστικές σακούλες και υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν 300 φορές περισσότερες σακούλες. Και αυτό το χάσμα είναι τεράστιο. Επομένως, κάποιες πολιτικές είναι ήδη πιο αποτελεσματικέ και κάποιες άλλες όχι. Το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει πλέον να εφαρμοστεί και να γίνει υποχρεωτικό μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στην πολιτική μου ομάδα ε, το θέμα ακόμα είναι υποσυζήτηση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Καταρχήν λοιπόν αυτό μας αποσχολεί και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, διαμορφώσουμε τις τροπολογίες μας. Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε την νομοθεσία απαγόρευση το 2020 είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θηλιάδος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κυρία Μίλλερ. Ή στον κύριο Μίλλερ. Α, η κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για τα έργα της και να ευχαριστήσουμε επίσης τους βουλευτές που είναι εδώ για ε, την συζήτηση. Εμείς θα λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα τα έχουμε υπόψη μας κατά την διαδικασία συνδιαλλαγής ή και συναπόφασης. Επιτρέψτε μου τώρα να εντάξουμε αυτή την πρόταση ε, στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλειών που εξελίσσονται. Γιατί όπως θα ξέρετε το πεδίο εφαρμογή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αλλά και οι συνομιλίες. Σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα όσον αφορά ε, το πόσο ρηπαίνουν αυτές οι πλαστικές σακούλες, οπότε και βέβαια υπάρχει θέμα με τα πλαστικά απόβλητα γενικότερα. Επομένως ε, είναι κάτω το ότι οι προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε πάνε πέρα οι πιο γενικότερες από αυτήν την πρόταση μου πολύ συγκεκριμένη γιατί εστιάζεται μόνο στο, στο, στα, στα, στη ρήπανση που προέρχεται από αυτές τις ε, ελαφρές ε, σακούλες τις λεπτές σακούλες. Θέλουμε επομένω, ε, και αυτό είναι η αφετηρία, το πώς δεν θα ρηπαίνεται η θάλασσα από αυτές τις πλαστικές σακούλες. Γιατί αυτές οι σακούλες ευθύνουν το 80% της ρήπανσης των ε, θαλασσών. Και επίσης αυτό το πλαστικό το 70% προέρχεται από ε, πλαστικά απόβλητα. Επομένως θα πρέπει να περιορίσουμε την ρήπανση από αυτές τις σακούλες και έτσι η μόνιση των θαλασσών θα μειωθεί. Έχει υπάρξει αίτημα του Συμβουλίου έχουν διατυπωθεί επίσης προς εμάς αιτήματα των ε, βουλευτών που και μας διαβιβάσετε, δηλαδή αιτήματα του κόσμου όσον αφορά το ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Γι' αυτό και έτσι και εμείς αρχίσαμε τις ενέργειες για να καταλήξουν σε αυτή την πρόταση και έτσι να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία ελπίζουμε ότι σύντομα θα εγκριθεί. Ούτως ώστε να μπορέσουν τα μέλη να προχωρήσουν στην λήψη μέτρων ε, που να εστιάζονται σε αυτό το πρόβλημα. Όμως, δεν έχουμε μόνο αυτό το πρόβλημα όσον αφορά τα απόβλητα και κυρίως τα πλαστικά που προέρχονται από συσκευασίε. Υπάρχουν ε, ταυτόχρονα τώρα σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές πρωτοβουλίες. Πρώτα πρώτα έχουμε την ευρεία ε, αναθεώρηση της οδηγίας για συσκευασία, ε, αυτό που λέμε fitness check και επίσης με τις σχετικές οδηγίες Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσον είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Μήπως είναι απειριχαιωμένες, άχρηστες οι διατάξεις αυτών των, ε, ε, των οδηγιών. Ιδίως ε, τις οδηγίες για τα απόβλητα και έτσι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες διατάξεις ώστε να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούμε. Ανακύκλωση, ποσοστό επαναχρησιμοποίησης μήπως και πρέπει να διαφοροποιήσουμε ανάλογα με το είδος των πλαστικών της ε, ρυθμίσεις μας. Επομένως, η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ε, αρκετά ευρία αυτή η διαδικασία και θεωρήσαμε ότι η μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών οδηγεί αυτή τη δραματική κατάσταση όσον αφορά τι θάλασσε. Και γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα πρέπει να, να καθυστερούμε. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό το fitness check και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει και άλλη μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία για τα πλαστικά απόβλητα γιατί θα πρέπει να έχουμε συντονισμένε προσπάθειε που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Επίσης υπάρχει μια πράσινη βίβλος που έχει δημοσιευθεί, υπάρχει επίσης ε, διαβούλευση, συζητήσεις, εξελίξει. οπότε και το αποτέλεσμα τέτοιων συζητήσεων και μελετών θα γίνουν και θα αναθεωρηθούν. Ως χρονοδιάγραμμα τώρα έχουμε πει ότι μέχρι το θέρος θα πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σαν αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό, για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτής της οδηγίας. Άρα μέχρι το 2015 δεν θα έχουμε κάποια αναθεώρηση της ισχύους οδηγίας. Το 2015-2016 και γι' αυτό ε, λέμε ότι τώρα ε, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το βελνικές αυτής της πρότασης. Δεν ρυθμίζονται εδώ διαφορετικά είδη πλαστικού. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ρήπανση από τις πλαστικές σακούλες. στην αγορά. Κυκλοφορούν δύο διασπόμενες σακούλες. Αλλά σε πάρα πολύ συγκεκριμένες ε, και ενδεχόμενες συνθήκες ε, μπορεί να γίνει κομποστοποίηση και βιοδιάσπαση ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία που προφανώς αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχουν στη θάλασσα οπότε ό,τι σακούλα πεταχτεί εκεί ό,τι είδου και να είναι, οξοδιασπόμενοι, διδιασπόμενοι παραδοσιακοί, όλες αυτές θα διαλυθούν σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια, μικρό κομματάκια, τα οποία πρόκειται να παραμείνουν στο περιβάλλον, όσο θα έμενε οποιοδήποτε είδος πλαστικού και γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν ασχολούμεθα με την βιοδιάσπαση κάτι άλλο ε, που αφορά αυτές τις πάρα πολύ ελαφρε και λεπτές σακούλες, αυτές που χρησιμοποιούμε για τα φρούτα και λαχανικά. Δεν εξαιρούνται και αυτές από την ε, ε, πρόταση οδηγίας. Το μελετήσαμε. Τελικά όμως αν πάτε στο σούπερ μάρκετ θα, θα δείτε σε ρολά αυτές τις σακούλες θα και παίρνετε όσες θέλετε. Και πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς να χρειάζεται. Γιατί ο κόσμος έχει αυτή τη συνήθεια να τις παίρνει. Measures like putting an indication above these rolls of plastic, please think of the environment. Take... Πότε λέμε να βάλουμε εκεί πέρα μια ταμπέλα που να λέει σκεφτείτε το περιβάλλον. Πάρτε μόνο ό,τι χρειάζεται και τα, τα κρατημέλη μπορούν να μειώσουν επομένω τη χρήση έτσι αυτών των ε, πλαστικών σαγούλων. Ο, λόγος που ακόμα καλύτερο είναι ότι θα ε, υπάρχει ακόμα περιθώριο να μειωθεί η χρήση και αυτών των ε, πλαστικών σαγούλων. Η δε πρόταση παραμένει τέτοιου γενικού είδους γιατί θεωρήσαμε ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να ορίσουν ειδικότερα για το, το πώς θα εφαρμόσουν τυχόν μέτρα. Επίσης, όπως έχει σήμερα η κατάσταση, ξεκάθαρα προκύπτει ότι η οδήποτε μέτρο που λαμβάνεται από κράτος μέλος έχει άμεσα αποτελέσματα σχεδόν. Και Προήψε ότι τα, τα, τα κράτη-μέλη υπάρχει υψηλό, υψηλός ρυθμός κατανάλωσης και άρα η επικουρικότητα εδώ ελήφθη υπόψη. Δηλαδή είναι υποχρεωμένα τα κρατημένα να ενεργήσουν, αλλά απόκειται σε εκείνα το πώς θα ενεργήσουν. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία τα οποία εθίξατε και σα ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε Ελπίζω κάποιος να έχει σημειώσει όλες τις παρεμβάσεις ε, για τον εισηγητή, γιατί ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Και λοιπόν θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων είναι η επόμενη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε λοιπόν νωρί νωρίς εκεί για να τις προλάβετε. Και λυπάμαι που σας το λέω εγώ, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να είναι σε μία γλώσσα μόνο λόγω χρόνου, έλλειψης χρόνου. Στα αγγλικά λοιπόν και ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος στα γαλλικά. Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα περνάμε στους ανεξελίξει τριημερή διαλόγου σε ό,τι αφορά το πακέτο επενδύσεων. Ο κ. Λάμπστορφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. έω τώρα έχει γίνει μία συνάντηση. Μία διαβούλευση σε πλαίσια τριμερούς ε, διαλόγου και θα πω ότι όλες οι διαπραγματεύσεις πήγαν πολύ καλά, όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν. Έγινε και ένα follow-up μετά τις τεχνικές συναντήσεις. Στην έκθεσή μου λοιπόν. Παρουσιάστηκαν δύο τεχνικές δυσκολίες οι οποίες και επιλύθηκαν. Άρα έως τώρα κανένα πρόβλημα θεωρώ ότι θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια και θα εγκριθεί. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εξαιρετική αυτή η αναφορά. Θέλει κανένας να κάνει κανένα σχολείο, καμία προσθήκη. Η σιωπή λοιπόν εκλαμβάνεται ως συνένεση. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να σας διευκρινίσω ότι η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στην... στο Στρασβούργο, Δευτέρα. Και νομίζω ότι είναι και η τελευταια τελευταία συνάντηση 17-18 Μαρτίου πριν τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση. τον κυριακό.